Ε, και κύριοι, ε, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία θα κάνω δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, η κυρία Ελένη Θεοχάρους ε, εγκατέλειψε την πολιτική ομάδα του ΕΛΚ και από την Δευτέρα Τρίτου